Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων θα ήθελα να καλωσορίσω την υποψηφία επίτροπο, την κυρία Βέρα Γιούροβα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον κύριο Μωράες, τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, την κυρία Βίκη Φόρντ, υπεύθυνη για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και η Ρατσέκ Γκαρσία Πέρες, πρόεδρο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων να καλωσορίσω τα μέλη όλων αυτών των επιτροπών που ε, συνδιοργανώνουν τη σημερινή ακρόαση. Η κυρία Γιούροβα, όπως και εγώ, είναι από την Τσεχία και γι' αυτό θα αποφύγω κάποια δυσθυμία, ίσως ε, λέγοντας ότι λέγεται Γιούροβα και όχι Τζούροβα, ούτε Ζούροβα αλλά Γιούροβα, Λοιπόν, θα εκτιμήσει την προσπάθεια που κάνω η υποψηφία επίτροπος νομίζω. Η κυρία Γιούροβα λοιπόν έχει ένα πολύ ευρύ ε, χαρτοφυλάκιο. Το πιο σημαντικό θέμα για μένα είναι το θέμα των αστικών υποθέσεων για το οποίο είναι υπεύθυνη η δική μου επιτροπή αναμένονται πολλές πρωτοβουλίες όπως ε, το σύστημα για τις ε, διασύνοριακές, ε, συστήματα, διασύνοριακά συστήματα πληρωμών. Ε, επίσης το θέμα του εταιρικού δικαίου είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με θέματα όπως η κοινωνική ευθύνη για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, υπό το φως ε, των κατευθυντηρίων γραμμών ε, για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλούμεθα να αξιολογήσουμε τους υποψηφίους επιτροπούς επί τη βάση των γενικών τους γνώσεων, της ευρωπαϊκής τους αποσίωσης και της προσωπικής τους ανεξαρτησίας. Αξιολογούμε επίσης και εκτιμούμε τις γνώσεις που έχουν για το χαρτοφυλάκιό τους, όπως επίσης και τις δυνατότητες επικοινωνίας που έχουν. Ε, μας ε, έδωσε γραπτές απαντήσεις στο πραπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο η υποψηφία επίτροπος. Ε, οι γραπτές απαντήσεις έχουν διανεμηθεί σε όλες τις γλώσσες τα μέλη των επιτροπών μας. Η διάρθρωση λοιπόν της συνάντησης θα είναι εξή. Θα κάνει μία παρουσίαση όχι άνω των 15 λεπτών η κυρία Γιούροβα. Θα έχει επίσης 5 λεπτά στο τέλος της συνεδρίασης για να κλείσει τη συζήτηση. Ε, και ο πρόεδρος θα έχει αυτή τη δυνατότητα αλλά για δίλεπτο. Μετά από τη εισαγωγή της κυρίας Γιούρεβα θα ακολουθήσουν 45 ερωτήσεις, ε, ένα λεπτό απάντησης ε, ή μάλλον ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Δεν υπάρχουν δυνατότητες συμπληρωματικών ερωτήσεων ή συστήματος catch θα ήθελα να ζητήσω από την υποψηφία επίτροπο και τους βουλευτές να σεβαστούν τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Συμφωνήθηκε ότι οι ερωτήσεις θα τεθούν ως εξής, με την εξής σειρά. Νομικές υποθέσεις πρώτα, δημόσιες ελευθερίες μετά, εσωτερική αγορά, και προστασία του καταναλωτή και τέλος ε, ε, Επιτροπή ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Έχουμε διερμηνία στη διάθεσή μας και οι ομιλητές μπορεί να χρησιμοποιούν την γλώσσα τους, αλλά καλούνται παρακαλώ να μην ομιλούν πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Μωράες. Point of order. Διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα. Ίσως υπάρχει παρεξήγηση από τη δική μου πλευρά. Αλλά για τη σοσιαλιστική ομάδα η προετοιμασία μας βασιζόταν στο ότι προηγούνται οι ερωτήσει τη Επιτροπή ΛΥΜΠΑ και μετά τη Νομική Επιτροπή. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι ποιο απόφασε, αποφάσισε να αλλάξει αυτή η σειρά και γιατί έχει αλλάξει και επί ποιας βάσης έχει αλλάξει. Uh, Χθε έλαβε χώρα μια συμφωνία για τη σειρά των ερωτήσεων, για τη σειρά των επιτροπών στην ε, υποβολή ερωτήσεων. Ε, πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων συγκεκριμένα. Κύριε Μωράης, λοιπόν, έχετε τρία λεπτά για την ενακτήρια σας ομιλία. Όχι. Εντάξει, θα δώσω τα 15 λεφτά στην κυρία Γιοούροβα. Έχετε το λόγο κυρία.